Η κυρία Πρόεδρος. Αρχίζει η συνεδρίαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης σας έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχουν, οπότε εγκρίνονται τα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής. Ε, και τώρα ερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη η οποία προβλέπει την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με το ρόλο του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών. Θα πάρουν το λόγο καταρχάς η κυρία Πακ, ως συντάκτης της ε, ερώτησης αυτής. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά κυρία Πακ